Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Μπορούμε να αρχίσουμε τις εργασίες μας. Thank you very much for taking... Σας ευχαριστώ πολύ που καθίσατε. την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και πριν ε, αρχίσουμε τις εργασίες μας, θα ήθελα οι διερμηνείς να μας παρουσιάσουν το μήνυμά τους, την δήλωσή τους όσον αφορά την απεργία τους. Παρακαλώ. Σήμερα είναι η 36η ημέρα της διαμαρτυρία μας κατά τη μονομερούς επιβολής άδικων συνθηκών εργασία για του διερμηνεί από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου. Με λύπη μας σας πληροφορούμε ότι δεν θα χορηγήσουμε καμία υπέρβαση ωραρίου. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. Ωραία, ευχαριστούμε. Τώρα συνεχίζουμε και να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη πρώτα απ' όλα. Έχετε την ημερήσια διάταξη. Σωστά, υπάρχουν σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις. Όχι από ό,τι βλέπω. Ωραία, οπότε δεχόμαστε ως έχει την ε, ημερήσια διάταξη. Ο ανακοινώσεις του Προεδρού. Δεν έχω τίποτα. Το μόνο είναι για την αντιπροσωπεία μας στην Ουάσιγκτον και τη Βοστόνη. Αλλά ο κύριο Ομαζέ θα μας ενημερώσει για την αποστολή αυτή μετά την ψηφοφορία, έτσι όχι τώρα. Μετά την ψηφοφορία. Ωραία. Οπότε συνεχίζουμε και περνάμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την ε, έκθεσή μας όθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συσηγητής μας είναι ο κύριος Χέτμαν. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ήταν 22 Μαΐου. Μας έφτασαν 137 τροπολογίες. Ο εισηγητής κατέληξε σε 23 συμβιβαστικές τροπολογίες. Έγιναν διαπραγματεύσεις μεταξύ των ομάδων και τώρα θα ψηφίσουμε. Κύριε Χέτμαν, θέλετε κάτι να πείτε πριν την ψηφοφορία? Όχι, ωραία. Οπότε αρχίζουμε την ψηφοφορία ευθύ αμέσως. Και αρχίζουμε με τη σεβαστική τροπολογία αριθμός 6. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, η τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά για την ε, τροπολογία 57. Τροπολογία 57. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Τώρα, συνεχίζουμε. Συμβιβαστική τροπολογία 12. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 69, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 70, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 81. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 87. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 88. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 89. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 90. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 102 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 103 υπέρ, κατά, Α, συγγνώμη, λέει πρόεδρο. Ναι, με προφορική τροποποίηση. Είναι κανεί κατά τη προφορική τροποποίηση, όχι. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 103 με την προφορική τροποποίηση. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 107. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 108. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 109. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 119. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 120. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 124 με προφορική τροποποίηση. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροποποίησης, όχι. Ψηφίζουμε την τροπολογία 124 λοιπόν με την προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 133 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 134, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 135, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 136, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 137 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στις τροπολογίες που προτείνει η Επιτροπή Πολιτισμού. Καλτ 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Καλτ 4, 41 και 3 καταπίπτουν εξαιτίας της συμβαστικής. Τώρα είμαστε στην 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Καλτ 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επόμενες καταπίπτουν. Καλτ 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Καλτ 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Καλτ 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλτ 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλτ 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Καλτ 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Καλτ 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Καλτ 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Καλτ 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Και εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Οπότε τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Τώρα, στην Επιτροπή μας και πάλι και στην ημερήσια διάταξη επιστρέφουμε με το επόμενο σημείο. Uh, Συνεχίζουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη. Το επόμενο σημείο είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Αλέξη Χαρίτσι. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομία και Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 2015 κάθετος 1839. Η Επιτροπή μας ενέκρινε έκθεση για ειδικά μέτρα όσον αφορά την Ελλάδα υπό τα πλαίσια του κανονισμού αυτού. Και αυτό στην προηγούμενη συνεδρίασή μας. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Αριμόντ, μας υπέβαλε και μας παρουσίασε την έκθεσή του. Συζητήσαμε λοιπόν την έκθεση αυτή στην Ολομέλεια και στη συζήτηση τα μέλη εξέφρασαν την επιθυμία να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον αρμόδιο υπουργό για αυτό το θέμα. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας που δέχτηκε την πρόσκλησή μας να έρθει εδώ σήμερα. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τις εθνικές αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνε για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Και αυτό είναι και το αντικείμενο της έκθεσής μας εξάλλου. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον Υπουργό για την παρουσίασή του πρώτα. Και μετά θα ζητήσουμε από τα μέλη της Επιτροπής μας να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους, τα σχόλιά τους με τον παραδοσιακό τρόπο. Αρχίζουμε με τους συντονιστές δηλαδή και μετά θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους βουλευτές της Επιτροπής μας. Οπότε κύριε Υπουργέ έχετε το λόγο. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ε, να ευχαριστήσω καταρχάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Ρέτζη και την Πρόεδρο ε, κυρία Μιχαήλοβα προσωπικά για την ε, πρόσκληση. Νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση ε, δεν θα μπορούσε να διεξάγεται σε πιο κατάλληλη συγκυρία με την έννοια ότι σε λίγες εβδομάδες η Ελλάδα εξέρχεται επιτυχώς από τα προγράμματα προσαρμογής ανακτώντας τον έλεγχο επί της πολιτικής της, τη δυνατότητα δηλαδή, αλλά και την ευθύνη να σχεδιάζει το μέλλον της και να συμμετέχει ισότιμα στις διεθνείς εξελίξεις. Καθοριστική σημασία για αυτή την εξέλιξη ήταν βεβαίω η συμφωνία για την διευθέτηση του χρέου στο τελευταίο Eurogroup τη 21η Ιουνίου, η οποία καθιστά βιώσιμο το ελληνικό χρέο σε μέσο πρόθεσμη βάση, μειώνει σημαντικά τι αιτήσει δαπάνε εξυπηρέτησή του και επιτρέπει στη χώρα να επανέλθει με ασφάλεια στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή η ελληνική οικονομία κινείται πλέον σταθερά με ρυθμούς ε, ανάπτυξης, 1,4% του ΑΕΠ πέρυσι το 2017. Ήταν η πρώτη χρονιά μετά από 10 χρόνια που είχαμε αύξηση του ΑΕΠ άνω του 1% και με τα μηνύματα για το 2018 να είναι ακόμα πιο ελπιδοφόρα, 2,3% αύξηση του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2018. Εξίσου σημαντικό όμως με την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ είναι το γεγονός ότι η βελτίωση αυτή των μακροοικονομικών μεγεθών εδράζεται σε σημαντικά ποιοτικά στοιχεία, όπως είναι η αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες έφτασαν στο 33% του ΑΕΠ το 2017, για πρώτη φορά σε αυτό το ποσοστό, η αύξηση των, της μεταποίησης και της βιομηχανίας κατά 4,5% την περασμένη χρονιά, το 2017 σχέση με το 2016 και η αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων κατά 29,5% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ενώ ταυτόχρονα έχει σημειωθεί μια σημαντική μείωση της ανεργίας, η οποία κινείται στο 20,1% από 27% που βρισκόταν πριν από τρία χρόνια. Ταυτόχρονα με αυτές τις θετικές εξελίξεις, η κυβέρνησή μας πήρε την πρωτοβουλία να εκπονήσει τη δική της αναπτυξιακή στρατηγική, με την οποία δεσμεύεται αφενός να διαφυλάξει την δημοσιονομική και μακροοικονομική σταθερότητα που με θυσίες κατέκτησε η χώρα τα τελευταία χρόνια, να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το οικονομικό περιβάλλον, διευκολύνουν τις επενδύσεις και θωρακίζουν την ανάπτυξη και να προχωρήσει στη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους με ποιοτικέ υπηρεσίες προς όλους τους πολίτες, αλλά και με μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων και τη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασία. Τέλο, και αυτό αποτελεί επίση μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μα, προχωρούμε στην επίλυση χρόνιων διπλωματικών προβλημάτων με γειτονικέ χώρε, όπω η πρόσφατη συμφωνία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία, συμβάλλοντα έτσι αποφασιστικά στη σταθερότητα, την ειρήνη και τη συνανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Με την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, θα έλεγα ότι κλείνει αυτός ο κύκλος της ευρωπαϊκής κρίσης που άνοιξε το 2009 και η οποία κρίση δοκίμασε τις αντοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης και αμφισβήτησε το μέλλον της. Η κρίση, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, βρήκε την Ευρωπαϊκή Ένωση απροετοίμαστη χωρί τα κατάλληλα εργαλεία και την αποφασιστική βούληση να δοθούν συνολικές λύσει σε προβλήματα που δεν ήταν μόνο εθνικά, αλλά πρωτίστως ευρωπαϊκά. Μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει δυστυχώ τον κανόνα σε αυτήν την ε, λογική υπήρξε η πολιτική συνοχή. Το βασικό εργαλείο που διαθέτει η Ένωση για την προώθηση τη σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών, τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και την καταπολέμηση της ανεργίας. Η πολιτική συνοχής λειτουργήσε και εξακολουθεί και σήμερα ακόμα να λειτουργεί ως το πραγματικό αντίβαρο στις φυγόκεντες τάσεις που έχει δημιουργήσει η κρίση. Για την Ελλάδα, η πόροι της πολιτικής συνοχής, οι πόροι των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ήταν ανέκαθεν πάρα πολύ σημαντικοί αποτέλεσαν για δεκαετίες τη βασική πηγή χρηματοδότησης μικρών και μεγάλων υποδομών σε όλη τη χώρα. Αλλά βεβαίως, ειδικά στα χρόνια της κρίσης, οι πόροι αυτοί υπήρξαν καθοριστικοί. Τα χρόνια αυτά η ελληνική οικονομία βίωσε μια πολύ μεγάλη κρίση από επένδυση και συνθήκες πιστοτική ασφυξίας. Οι επενδύσει μειώθηκαν δραστικά τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Αναγνωρίζοντα λοιπόν την σημασία που έχουν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ειδικά μέσα στην κρίση, η κυβέρνησή μα έκανε έναν αγώνα δρόμου τα τελευταία τρία χρόνια, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκεί που θα έχουν το μεγαλύτερο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία μπορούμε ευθαρσώς να πούμε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι κράτησαν κυριολεκτικά την ελληνική οικονομία όρθια. Χρηματοδότησαν κρίσιμα έργα υποδομών, προγράμματα για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετώπισαν τεράστια έλλειψη ρευστότητα. Θεωρούμε ότι η προσπάθεια την οποία κάναμε έφερε απτά αποτελέσματα. Η Ελλάδα αξιοποίησε πλήρως τους πόρους της προγραμματικής περίοδου 2007-2013 δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Ενεργοποίησε πρώτη τα προγράμματα της νέας περίοδου 2014-2020 και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την ίδια στιγμή, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, η χώρα μας βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης ανά ε, κατακεφαλήν ΑΕΠ και στην αξιοποίηση των πόρων του άλλου μεγάλου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου, του Σιδίου Juncker. Ενώ συνεργαζόμαστε στενά με τους μεγάλους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, διασφαλίζοντας πρόσθετα κονδύλια για την ελληνική οικονομία. Σε όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, πολύτιμος αρρωγός στάθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μα χαροποιεί το γεγονός ότι στο τελευταίο διάστημα και με δημόσιες τοποθετήσεις Εξωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζουν αυτά τα πολύ θετικά αποτελέσματα. Σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν το 2015, όπως η χρηματοδότηση κατά 100%, υπήρξαν καθοριστικά ώστε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε έγκαιρα όλους τους πόρους της περίοδου 2007-2013 και να ολοκληρώσουμε κρίσιμα έργα όπως για παράδειγμα οι μεγάλοι εθνικοί αυτοκινητόδρομοι που πολύ πρόσφατα ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε κυκλοφορία. Η δε αύξηση της προκαταβολής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 που επίσης ε, αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια περίοδο, μας έδωσε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε τάχιστα τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περίοδου και να έχουμε, όπως είπα και πριν, αυτή τη μεγάλη απορρόφηση που παρουσιάζεται σήμερα και πιστέψτε με αυτά δεν αποτελούν αν θέλετε απλούς δείκτες ή αφηρημένους ε, αριθμούς και νούμερα. Οι πόροι αυτοί μετουσιώθηκαν σε πολύτιμα έργα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, σε κρίσιμες υποδομές που χρόνιζαν εδώ και δεκαετίες, αλλά και σε σημαντικές νέες θέσεις εργασίας που συνετέλεσαν έτσι ώστε να μειωθεί αυτό το εξωπραγματικό ποσοστό ανεργίας το οποίο ε, υπήρχε στη χώρα πριν από λίγα χρόνια. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε ε, όσο πιο συνοπτικά μπορώ να παραθέσω μερικά συγκεκριμένα στοιχεία για να δείξω τις θετικές επιπτώσεις από την αλλαγή του κανονισμού. Η άμεση καταρχάς επίπτωση στη διαθέσιμη ρευστότητα ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2015 και 468 εκατομμύρια ευρώ το 2016 άμεσα με την ενεργοποίηση του νέου κανονισμού, δηλαδή συνολικά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ τα οποία βοήθησαν ώστε οι συνολικές πληρωμές του κεντρικού λογαριασμού των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για το 2015 και το 2016 να ανέλθουν σε 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πόροι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για την ασφαλή, αποτελεσματική και αποδοτική ολοκλήρωση των έργων όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Εκτός βεβαίως των άμεσων ε, επιπτώσεων, δημοσιονομικών επιπτώσεων, υπήρξαν και έμεσε συνέπειες από την κινητοποίηση της οικονομίας, τις πληρωμές ολοκλήρωσης έργων, τη μείωση της ανεργία και την αύξηση των εισοδημάτων. Αυτές οι έμεσε επιπτώσεις μπορούν να εντοπιστούν στα στοιχεία της φοροδοτικής ικανότητας της οικονομίας. Το γεγονό δηλαδή ότι για το 2016 είχαμε μια αύξηση φορολογικών εσόδων κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2015 και αυτό ήταν μια εξέλιξη η οποία εμέσως συνδέεται και με την ε, ορθή ε, εκτέλεση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά την επίπτωση στην ανάπτυξη και με χρήση του πολλαπλασιαστή που χρησιμοποιείται για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις ex post αξιολογήσεις που κάναμε για την περίοδο 2007-2013, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ επενδύσεις της πολιτικής συνοχής, για αυτήν την προγραμματική περίοδο 7-13 παράγονται 2,74 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετου ΑΕΠ για την ελληνική οικονομία μέχρι και το 2023. Το να εκτιμηθούν οι ποιοτικέ επιπτώσεις ε, ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής του κανονισμού είναι βεβαίως αντικειμενικά και επιστημονικά ε, πολύ δύσκολο. Είναι όμως σημαντικό να τονίσουμε ότι η θετική επίπτωση της πολιτικής συνοχής συνολικά, άρα και της βελτίωσης του κανονισμού για την Ελλάδα, είναι ορατή στο οικονομικό και κοινωνικό γύρνεσθε της χώρας και των περιφερειών της. Ορισμένα λοιπόν ποιοτικά σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Επιτεύγματα της, περίοδου, της προγραμματικής περίοδου λοιπόν 713, νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης περίπου 27.000, εκ των οποίων 23.000 σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 3.500 σε νέους ερευνητές. 255.000 άνεργοι που επωφελήθηκαν από προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Ενίσχυση 40.000 περίπου επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Περισσότερο από 3.500 χιλιόμετρα οδικών αξώνων κατασκευάστηκαν ή βελτιώθηκαν με την χρήση των προγραμμάτων αυτών, ενώ και περισσότερα από 160.000 άτομα ευπαθών ομάδων από δράσει κοινωνική ένταξη ωφελήθηκαν από αυτά τα προγράμματα. Αυτά για την περίοδο 7-13. Σε σχέση με τη νέα προγραμματική περίοδο, την περίοδο 14-20, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουν ήδη δημοσιευθεί προσκλήσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη λοιπόν προγράμματα συνολικού ε, προπολογισμού 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή περίπου το 76% του συνόλου των διαθέσιμων πόρων έχει ήδη ενεργοποιηθεί, ενώ οι πραγματοποιηθήσεις, οι ήδη σε συνολικές δαπάνες ανέρχονται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά στι κορυφαίε θέσει μεταξύ των κρατών μελών στην απορρόφηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, του ΕΣΠΑ 1420. Κατά την εκτίμησή μα, ο στόχο, ο οποίο έχει τεθεί από τον κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ΝΙΣΙΝ 3, είναι ένα στόχο απόλυτα εφικτό και αποτελεί βεβαιότητα για την Ελλάδα ότι κανένα επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν κινδυνεύει από απώλεια πόρων για τα έτη 2018 και 2019 η ενεργοποίηση όλων αυτών των προγραμμάτων μας έδωσε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στη δημιουργία κάποιων εμβληματικών δράσεων. Θα αναφέρω συνοπτικά κάποιες από αυτές, απλά για να έχετε μία ε, γενική εικόνα. Συστήσαμε λοιπόν ένα νέο Ταμείο Υποδομών με δημόσια δαπάνη 450 εκατομμύρια ευρώ με σκοπό να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων υποδομής με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης. Δημιουργήσαμε επίσης το Ταμείο Επιχειρηματικότητας 2 με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 400 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο χορηγεί δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συστήσαμε σε συνεργασία με το EIF, το European Investment Fund, το νέο Ταμείο Equifund, Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, το οποίο σύμφωνα με, την, το EAF ε, είναι το μεγαλύτερο αντίστοιχο Ταμείο Equity Funding, το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται ε, σε χώρα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ υλοποιούμε και πολλά σημαντικά έργα ε, ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, Διπλασιάσαμε μάλιστα του σχετικού σχετικούς πόρους λόγω τη πολύ μεγάλη ζήτηση που παρουσιάζεται σε σχέση με την ε, εξοικονόμηση ενέργεια σε κατοικίε. Ταυτόχρονα, επειδή το ζήτημα της έρευνα και της σύνδεση της έρευνα με την πραγματική οικονομία είναι πάρα πολύ κρίσιμο, υλοποιούμε την πιο εμβληματική, θα έλεγα, δράση του νέου ΕΣΠΑ, που είναι το πρόγραμμα που ονομάζεται Ερευνό Δημιουργό Καινοτομό, που έχει ακριβώ ω στόχο με έναν πολύ σημαντικό προπολογισμό 410 εκατομμυρίων ευρώ να ενισχύσει τη σύνδεση των ερευνητικών ιδρυμάτων με την πραγματική οικονομία, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περισσότερες από 4.000 νέες ποιοτικέ θέσεις εργασίας για ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό θα δημιουργηθούν από αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Ενώ και πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν είχαν υλοποιηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες, υλοποιούνται τώρα μέσα από τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως είναι για παράδειγμα το έργο του κτηματολογίου, η προμήθεια μέσων δίωξης για τις τελωνιακές υπηρεσίες και άλλες βασικές υποδομές μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ε, δικτύων. Σε ό,τι αφορά τέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της περίοδου 2014-2020 και με δεδομένη την ανάγκη αδιάλειπτης παρουσίας δράσεων ανάσχεση ανεργία και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, υλοποιούνται μια σειρά από δράσεις, όπως πρωτοβουλίες για την απασχόληση των νέων, τα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση του κοινοφελούς εργασίας, η συνέχιση επιτυχημένων προγραμμάτων, όπως είναι τα προγράμματα για τους βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμού, αλλά και τα κέντρα κοινότητα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχεια. Συνολικά, ε, πέρα από τα επιμέρους προγράμματα ε, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό και δώσαμε ιδιαίτερο βάρος εκεί τα τελευταία χρόνια, είναι το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε θεσμική αναβάθμιση στις υπηρεσίες οι οποίες ε, είναι επιφορτισμένες με την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, με την ενίσχυση της διαχειριστικής του επάρκειας, αλλά και τη δημιουργία θεσμικής μνήμης στην ελληνική δημόσια διοίκηση που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Με βάση όλα τα παραπάνω και τις ε, επιτυχίες που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις Γενικές Διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιες για την πολιτική συνοχή, όπως επίσης και την Επιτροπή για την πρόταση η οποία πρόσφατα κατατέθηκε για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 η οποία προβλέπει αύξηση των πόρων για την Ελλάδα κατά 8%. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα ε, γενικότερο σχόλιο. Αυτή την περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητιέται ο προπολογισμό τη Ένωση για τα επόμενα χρόνια. Είναι μια συζήτηση που αφορά το μέλλον τη Ευρώπη. Τα διλήμματα που έχουμε να ε, αντιμετωπίσουμε, που μπαίνουν μπροστά μα, είναι επιτακτικά. Θα κινηθούμε πιο αποφασιστικά στην κατεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Ενωποίηση και θα αναπτύξουμε τα κατάλληλα εργαλεία που υπηρετούν αυτή την κατεύθυνση ή θα σταθούμε αμέτωχοι μπροστά στην άνοδο ευρωσκεπτικιστικών και εθνικιστικών δυνάμεων που θέτουν σε αμφισβήτηση την κοινή μας πορεία. Θα απαντήσουμε στις προσκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, στις προκλήσεις παγκοσμιοποίησης θέτοντας στο επίκεντρο των κοινών μας πολιτικών τις ανθρώπινες και τις κοινωνικές ανάγκες ή θα αφήσουμε τις περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές πολλές φορές ανισότητες να αποδυναμώσουν την κοινωνική συνοχή και να ροκανίσουν την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στο όραμα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης θα αντιμετωπίσουμε εν τέλει τις αυξημένες προσφυγικές ροές με επίκεντρο τις ευρωπαϊκές αξίες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης ή θα επιτρέψουμε λογικές εθνικής αναδίπλωσης ξενοφοβικών και μυσαλόδοξων φωνών να επικρατήσουν. Σε αυτή τη σύνθετη και γεμάτη προκλήσεις πραγματικότητα, επιτρέψτε μου να πω ότι η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει την καλύτερη εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσαρκώνει τι αξίε της αλληλεγγύη, της βιώσιμη και χωρί αποκλεισμού ανάπτυξη και τη κοινωνική συνοχής. Η ενίσχυσή της, λοιπόν, κατά τη γνώμη μα αποτελεί όρο ύπαρξη για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δοκιμάστηκε σκληρά τα τελευταία 8 χρόνια, τα χρόνια της κρίσης. Ε, αλλά βεβαίως, ε, μαζί με την οικονομική κρίση, κλήθηκε να αντιμετωπίσει και το βάρος των αυξημένων προσφυγικών ροών. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μέσα από την πολιτική της συνοχής επέτρεψε να μετριάσει η Ελλάδα τις συνέπειες αυτής της κρίσης, αλλά και να διαχειριστεί με ανθρωπισμό και αξιοπρέπεια την ε, ανθρωπιστική κρίση που δημιουργήθηκε στο προσφυγικό. Θα έλεγα λοιπόν, κλείνοντας, ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της συνοχής από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με τη δική σας βεβαίως πολύτιμη υποστήριξη, είναι το καλύτερο επιχείρημα για την ανάγκη ενίσχυση τη πολιτική συνοχή και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Σα ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας, γεμάτη στοιχεία. Γνωρίζετε ότι η δική μας Επιτροπή υποστήριξε τα έκτακτα μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα τα αποφασίζαμε πιστεύοντας ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να συνέλθει από την κρίση και να επιτύχει τα αποτελέσματα στα οποία αναφερθήκατε. Έχουμε το μόνιμο εισηγητή για την Ελλάδα, ο εισηγητής μας ε, και για την τελευταία έκθεση. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν. Μας έδωσε ένα πολύ θετικό μήνυμα για πολύ καλά αποτελέσματα. και ταυτόχρονα συμβούλεψε τις αρχές ε, της Ελλάδας να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστούμε λοιπόν για την ενημέρωση και για τα μελλοντικά βήματα στα οποία αναφερθήκατε και δίνω τώρα το λόγο στους ε, συντονιστές των πολιτικών ομάδων αν θέλουν να πάρουν το λόγο, όχι. Πολύ ωραία. Ο κύριος Σαριμό, μόνιμος εισηγητής μας για την Ελλάδα. Μπορείτε να... Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Υπουργέ. επεξεργαστήκαμε την έκθεσή μου με μια πολύ θετική νότα σε ό,τι αφορά τα έκτακτα μέτρα. Και παρακολουθήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία, επισκεφθήκαμε και επιτόπου την χώρα, συναντηθήκαμε με μέλη της κυβερνήσεως, με σημαντικούς φορείς της οικονομίας και σε όλη αυτή τη διάρκεια από το 2015 είχαμε πάντοτε την αίσθηση ότι τα λαμβάνουν σοβαρά τα πράγματα αυτά στην Ελλάδα και ότι προσπαθούν με ιδιαίτερα φιλόδοξο τρόπο να υλοποιήσουν τα έκτακτα μέτρα. Η συνεργασία μεταξύ της ελληνικής κυβερνήσεως και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα και νομίζω ήταν λίγο και το κλειδί για την επιτυχία, ότι δηλαδή τα κονδύλια αυτά έγιναν αντικείμενο μιας λογικής διαχείρισης και ότι μπόρεσαν τελικώς να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά. Κάτι που πιθανότατα δεν θα είχε γίνει αν δεν είχαμε αυτά τα specific measures, αν δεν τα είχαμε εγκρίνει αυτά και τα μέτρα για την συγχρηματοδότηση. Επιτρέψτε μου δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις για τα έκτακτα αυτά μέτρα και για τα έργα. Και ήταν λίγο και αυτό που ε, μας προκάλεσε κάποιες δυσκολίες ε, στην σύνταξη της εκθέσεως. Λάβαμε πάρα πολλά νούμερα σχετικά με ολοκλήρωση έργων. Αυτό καταρχήν είναι μια θετική είδηση. Μας έλειψε λίγο η απάντηση στο ερώτημα. Αυτά τα περίπου 150 priority project οδήγησαν πραγματι Μπορεί να το αποδείξει κανείς δηλαδή, μπορεί να το μετρήσει σε οικονομική ανάπτυξη. Εδώ, κατά την άποψή μου, λάβαμε κάπω λίγε πληροφορίε από την ελληνική κυβέρνηση, το ίδιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ερώτηση λοιπόν είναι, μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να μα δώσει αντικειμενικά μετρήσιμου δείκτε που να δείχνουν ότι ας πούμε η περιφερειακή πολιτική έχει ενισχυθεί και ότι γίνεται και αντιληπτή ως ενισχυμένη. Και δεύτερη ερώτηση τώρα που συνδέεται. Η ελληνική κυβέρνηση έχει φροντίσει ώστε αυτή η ολοκλήρωση των έργων προτεραιότητας να εμφανιστούν και στα μάτια του κοινού ως ευρωπαϊκά έργα. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν, ας πούμε, στους νέους αυτοκινητοδρόμους, γνωρίζουν ότι κυκλοφορούν σε αυτοκινητοδρόμους οι οποίοι κατά μεγάλο μέρος έχουν συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά χρήματα και προκαλείται μια πιο θετική εικόνα έτσι τη περιφερειακή πολιτική και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι θα αντιληφθεί ο κόσμο τότε ότι χωρί τα ευρωπαϊκά χρήματα δεν θα είχαν υπάρξει αυτά τα έργα. Και εδώ συνδέω και την διαρκή μα το διαρκές μας αίτημα, δηλαδή περιφερειακή πολιτική να είναι και προώθηση τη ευρωπαϊκή ιδέα. Γιατί είναι και καλύτερη διαφήμιση που μπορούμε να κάνουμε όταν δείχνουμε δηλαδή ότι τα ευρωπαϊκά χρήματα μπορούν να ωφελήσουν άμεσα τον κόσμο, του ανθρώπου. Εξού λοιπόν και θέτω την ερώτηση. Το γνωρίζουν οι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very... Ευχαριστούμε πολύ εκ τη ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών. Η κυρία Μπρέσο ή εσεί, η κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. πολύ σημαντικό για μας ε, το ότι μαθαίνουμε ότι οι πόροι της πολιτικής συνοχής δεν χρησιμεύσαν μόνο στη φυσιολογική φάση της πρόοδου της οικονομίας και της αναπτυξιακής πολιτικής αλλά χρησιμεύσαν και για παρεμβάσεις ε, σε τέτοιες περιπτώσεις ιδιαίτερα δραματικές. Σας συγχαίρουμε λοιπόν για τα αποτελέσματα που όπως φαίνεται είναι πολύ σημαντικά. Ακούγοντάς σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορείτε να μας βοηθήσετε να αξιολογήσουμε τι προγραμματισμός θα ακολουθήσει. Κατά την άποψή σας πιο συγκεκριμένα, η σύνδεση μεταξύ της πολιτικής συνοχής σε όλες τις τις πτυχές Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης, ε, ε, Κοινωνικό Ταμείο κτλ. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και οι συστάσεις ε, αναχώρα. Λειτουργεί, μπορεί να λειτουργήσει. Υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν υπερβολικές αναφορές σε προγράμματα πολιτικής συνοχής, ευρωπαϊκό εξάμεινο, συστάσεις Πώς ε, βλέπετε να γίνεται ο συντονισμός μεταξύ όλων αυτών των ε, ονομασιών προγραμμάτων, όλων αυτών των προγραμμάτων και ειδικότερα όσον αφορά το κοινωνικό ταμείο. Εσείς ε, πώς αξιολογείτε το συντονισμό μεταξύ κοινωνικού ταμείου και πολιτικής συνοχής. Για σας λειτουργήσε η παρέμβαση του κοινωνικού ταμείου σε συντονισμό με το νέο ευρωπαϊκό πυλώνα των ε, κοινωνικών δικαιωμάτων. Θεωρείτε μήπως ότι πρέπει να αλλάξει λίγο ή θεωρείτε ότι σε τελική ανάλυση η προηγούμενη δομή μπορεί να λειτουργήσει. Με ενδιαφέρει δηλαδή να καταλάβω στις τροποποίησεις που προτείνονται εσείς ως διαχειριστής ε, ε απευθείας διαχειριστής των ταμείων πώς τα αξιολογείτε τι συμβουλές θα δίνατε απλούστευσης ή τροποποίησης των κανονισμών. Τι θα προτείνατε. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε τώρα κύριε Τόμασιτς. Κύριε Τόμασιτς, όχι. Κύριε Βαρμιλτεμπορκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ και ευχαριστούμε για όλες τις εξηγήσει. Συγχαρητήρια στις προσπάθειες σας. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει μείνει είναι ακόμα λίγο πίσω αλλά συνέρχεται από την κρίση. Απομένουν πολλά να γίνουν. Πέρυσι, τον Ιούλιο του 2017, ε, είδαμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σταθερότητα ότι η Ελλάδα είχε μείνει πίσω και απήχε πολύ σε θέματα αποτελεσματικότητας και διακυβέρνησης. Και παραθέτω, εδώ λέγεται ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι πιο ελκυστικό μέρος επενδύσεων και χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για να ενισχυθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον. Κάποια παραδείγματα που αναφέρονται αναφέρουν για παράδειγμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ακαμψία σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς, αδικαιολόγητη και δυσανάλογοι περιορισμοί σε κάποια επαγγέλματα που δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί. Εξακολουθεί να πρέπει να εξυγχρονιστεί το πλαίσιο τη χρήση γη, βελτίωση τη αποτελεσματικότητα των μεταφορικών δικτύων και θα μπορούσα να συνεχίζω να μιλάω για αρκετά λεπτά. Υπάρχουν πολλά λοιπόν που πρέπει να γίνουν. Να το συνοψίσω με τρει λέξει. Μεταρρυθμίσει, μεταρρυθμίσει, μεταρρυθμίσει. Πρέπει να κάνετε, πιστεύω, ακόμα διαρθωτικέ μεταρρυθμίσει στη χώρα σα. Και φυσικά η Ευρώπη μπορεί να σα βοηθήσει διότι έχουμε εμεί το πρόγραμμα στήριξη των διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και η ερώτησή μου είναι πώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Κομισιόν και ειδικότερα τα προγράμματα διορθωτικών μεταρρυθμίσεων. ποιε είναι οι προτεραιότητές σας για τα επόμενα χρόνια, τι είδου μεταρρυθμίσει θα θέλατε να εφαρμόσετε κατά προτεραιότητα και ειδικότερα πώς αυτό αποτυπώνεται ε, στο πρόγραμμά σας ε, ανάπτυξης που παρουσιάσετε στο Eurogroup τον Απρίλιο φέτος που επίσης αποτέλεσε το αντικείμενο επίκρισης διότι παρουσιάστηκε και κλεισμένο το θυρών και για μας. Ξέρετε είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι ακριβώς βρισκόταν μέσα σε αυτή τη στρατηγική. Μπορείτε να μας πείτε τη σκέψη σας για τη στρατηγική αυτή και για τη σχέση με τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να καταλάβουμε τι θα γίνει και στο μέλλον διότι φυσικά απομένουν πολλά να γίνουν όπως είπα στην αρχή της παρέμβασή μου αλλά φυσικά μπορείτε να υπολογίζετε στη βοήθειά μας και τη επιτροπή αυτή, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα θα τα πάει καλύτερα στο εγγυσμένο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βανίστελμποργκ. Ο κύριο Παπαδημούλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, όσα μας παρουσίασε ο κύριος Χαρίτσης νομίζω ότι περιγράφουν μία ιστορία επιτυχίας στην οποία συμβάλαμε ιδιαίτερα ως Ευρωκοινοβούλιο μαζί και με την Κομισιόν και μαζί και με τις ελληνικές αρχές. Πριν από σχεδόν τρία χρόνια, το φθινόπωρο του 2015, μετά από πρόταση της Κομισιόν και έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα ποσοστό της τάξης του 90%, αποφασίσαμε την αλλαγή με τον κανονισμό 1839 του 2015. Μια εξαιρετική ρύθμιση. Μια ρύθμιση κατεξαίρεση για την Ελλάδα. Και τώρα βλέπουμε ότι οι καρποί αυτής της ρύθμισης λειτουργήσαν πολύ θετικά και για την Ελλάδα και για τις πολιτικές συνοχής και για την προώθηση της ιδέας ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα απέναντι στους ακροδεξιούς λαϊκιστές που ισχυρίζονται ότι πρέπει να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταργηθεί η πολιτική συνοχή. Και αυτή η αλλαγή δεν επιβάρυνε ούτε ένα ευρώ τους Ευρωπαίους φορολογουμένους. Το αποτέλεσμα ήταν δημοσιονομικά ουδέτερο. Απλώς έγινε μια πιο έμπροστοβαρής ρύθμιση για τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων. Και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος που αποτυπώνεται αυτή η αξιολόγηση είναι η έκθεση αριμών, την οποία πριν λίγες ημέρες εγκρίναμε με 36 υπέρ έναντι δύο μόνο που δεν ψήφισαν θετικά. Δηλαδή το σύνολο σχεδόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής. Νομίζω ότι κύριε Χαρίτσι, θα πρέπει να λογαριάζετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα αυτή την Επιτροπή ως σταθερό σύμμαχο και υποστηριχτή των προσπαθειών για ισχυροποίηση της πολιτικής συνοχής και για τις προσπάθειες που κάνει η χώρα μας, η Ελλάδα, να προχωρήσει το δρόμο των μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητες έτσι ώστε να μην ξαναχρειαστεί ποτέ η Ελλάδα να έχει είτε μνημόνια είτε εξαιρετικέ ρυθμίσει όπως ο κανονισμός 1839. Ε, και θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά στον κύριο Βαν Μίτεμπερκ. Είμαι βέβαιος ότι ο Υπουργός θα αναφέρει πολύ περισσότερα. Πριν τρία χρόνια οι δασικοί χάρτες στην Ελλάδα βρισκόντουσαν στο 0,6%. Το κτηματολόγιο, το Land Register, ήταν περίπου μια υπόθεση σχεδόν στο 0% τώρα προχωράει με ικανοποιητικού ρυθμού. βρίσκεται στο 30% και σύμφωνα με την Κομισιόν θα ολοκληρωθεί το 2021. Επομένω, ο στόχος της χώρας μου και των αρχών τη είναι να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να γίνει μια χώρα με ισχυρή διοίκηση, πιο φιλική στις επενδύσεις για να μπορέσει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της ε, πλεονεκτήματα. Η έξοδος από τα μνημόνια δεν σημαίνει σταματάμε τις μεταρρυθμίσεις, απορρίπτουμε την επιστροφή στο παλιό μοντέλο που γεννούσε ελλείμματα και χρέη με πολύ πελατειακό κράτος, πολύ φοροδιαφυγή, πολύ διαφθορά και θέλουμε να, η Ελλάδα να αξιοποιήσει με μοντέρνες μεταρρυθμίσεις όλες τα συγκριτικά πλονεκτήματα. Κύριε Βαν Μίλτερμπερκ, σας παραπέμπω στην έκθεση του ΟΣΑ, την πολύ πρόσφατη, και στην ομιλία του κυρίου Γκουρία, που λέει ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είναι πρώτη στη λίστα των δομικών ε, μεταρρυθμίσεων. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά νομίζω ότι όλοι μας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο που συμβάλαμε σε αυτό θα πρέπει να νιώθουμε ικανοποίηση γιατί η Ελλάδα σήμερα επιστρέφει και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν μερικά χρόνια. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ms. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το λόγο, κύριε Χένκελ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπουμε εδώ. Λοιπόν, ακούγοντάς σας, σκεφτόμουν ότι όλοι είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που ξαναμπαίνει στο δρόμο η Ελλάδα. Ε, συγχρόνως όταν κοιτάω τι γίνεται με την ανεργία των νέων, με την ένδια, πραγματικά δεν καταφέρνω να είμαι πλήρως ικανοποιημένη από την κατάσταση. Και αυτό πρέπει να υποθεί επίσης ότι μένουν πολλά ακόμα να γίνουν γιατί η κατάσταση, τουλάχιστον για κάποιες ε, ομάδες πληθυσμού, είναι πολύ δύσκολη. Τώρα, εγώ ε, θα διαφέρω από τους υπόλοιπους, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι είναι οι μεταρρυθμίσεις που θέλουμε τώρα πέρα από τόσα έχουν γίνει, γιατί όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, τα διάφορα προγράμματα, μεταρρυθμίσεις κτλ. έγιναν η προτεραιότητα για την επόμενη προγραμματική περίοδο, για την ε, συνοχή, για παράδειγμα. Οπότε το θέμα δεν είναι να κάνουμε μεταρρυθμίσει για τις μεταρρυθμίσει, είναι να δούμε πώς βάζουμε τι προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων αυτών. Γιατί χρησιμοποιήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις για πολλά πράγματα, μερικές φορές σε βάρος της καλής λειτουργίας της δημόσιας δίκησης, για παράδειγμα. Γιατί το να κόβουμε θέσεις απασχόλησης στο δημόσιο τομέα δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα γίνεται και πιο αποτελεσματικός, ότι θα υπάρχει ένα καλύτερο φορολογικό σύστημα ή ότι θα ελέγχεται αυτό καλύτερα. Όχι. Οπότε εσείς στα προγράμματα τα οποία ελοπείτε στην Ελλάδα, πώς θα θέσετε τις προτεραιότητες. Και σε μας τι θα λέγατε σαν συμβουλή από την εμπειρία που έχετε εσείς όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί υπάρχουν και άλλες χώρες που θα θέλανε ίσως να υλοποιήσουν τέτοια μέτρα και καλό θα ήταν να έχουν ακούσει τις δικές σας εμπειρίες από την Ελλάδα. Και πώς συνδέονται αυτά με τη χρήση των κονδυλίων συνοχής. Γιατί αυτό βρίσκεται στην καρδιά της κατανόησης για να καταλάβει κανείς πώς μπορεί να βοηθήσει τις ερθρωτικές μεταρρυθμίσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να πείτε περισσότερα γι' αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Σπυράκη είναι επόμενο μιλήτρια. Thank you, Madam Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μα. Είναι αναμφισβήτητο ότι η τροποποίηση του κανονισμού 1839 που έδωσε την εξαίρεση στην Ελλάδα που επέτρεψε δηλαδή να μην υπάρχει εθνική συμμετοχή για το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2007-2014 και έδωσε τη δυνατότητα υψηλής εμπροστοβαρούς χρηματοδότησης για το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2014-2020 ήταν η έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγγύης των εταίρων προς την πατρίδα μας η οποία βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και φαίνεται πως η απόδειξη αυτής της αλληλεγγύης διοχέτευσε πράγματι χρήματα στην Ελλάδα ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να πάρει ανάσα. Στην πραγματική οικονομία όμως, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να σας θέσω κάποια ερωτήματα και θα ήθελα πολύ καλόπιστα τις απαντήσεις σας. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα cohesiondata.eceuropa.eu/overview, η Ελλάδα φαίνεται να έχει για την περίοδο 2014-2020 δώσει στην πραγματική οικονομία μόνο το 17% των δυνατοτήτων της. Το 17% των δυνατοτήτων αυτού του κοινοτικού πλαισίου. Πρόκειται για τις δαπάνες και όχι για τις δεσμεύσεις. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι θέλω να μας πείτε πώς εξηγείται το γεγονός ότι ενώ υπάρχουν δεσμεύσεις δεν διοχετεύονται τα πραγματικά ποσά στην ελληνική οικονομία. Και για να γίνω ακόμα πιο ειδική σε αυτό. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η βάση της ιστοσελίδας που συγκεντρώνονται στοιχεία για όλα τα κράτη μέλη η ελλάδα δεν έχει ενισχύσει καμία μικρομεσαία επιχείρηση. είναι στη διάθεσή σας τα στοιχεία αυτά και μπορώ να σας τα δώσω και επειδή πραγματικά σας ρωτάω καλόπιστα μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν εισπράξει κάποια επιδότηση την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και γιατί αυτές δεν αναγράφονται στα επίσημα στοιχεία της κομισιόν. το τρίτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι πόσα νέα έργα χρηματοδοτήθηκαν από την εμπροσοβαρή χρηματοδότηση την περίοδο 15-16 και πόσα έργα ήταν έργα της προηγούμενης περίοδου, δηλαδή ήταν έργα phasing. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω τις απαντήσεις σας. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μονσκούρ. Yes. Έχετε το λόγο. Yes, Εκτός μικροφώνου, κύριε ομιλητής. Η προσοχή είχε δοθεί για πολύ καιρό στη χώρα σας, το ίδιο και στις κυβερνήσεις σας. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για ορισμένους, μάλιστα επίσης, ε, καταδείχθηκε ως υπεύθυνη για την καταστροφική κατάσταση στην οποία βρέθηκε η Ελλάδα. Σήμερα είμαστε ευτυχείς που έρχεστε να μας δείτε και να μας πείτε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί και κατά πολύ μάλιστα έχει μειωθεί η ανεργία, το ανάπτυξη έχει θετικό δείκτη, όλοι οι δείκτες φαίνεται είναι θετικοί. Συγχαρητήρια. Έχω δύο ερωτήσεις. Οι Έλληνες έχουν αντιλήψει του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ε, επανόρθωση της χώρας σας. Εσείς, ε, οι πολιτικοί, ως ε, υπεύθυνοι για τα περιφερειακά προγράμματα, έχετε την αίσθηση ότι κάνετε ό,τι πρέπει για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους λαούς και ειδικότερα στο δικό σας, να αποκατασταθεί η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο λαό σας. Μου φαίνεται σημαντικό για τις εποχές τόσο δύσκολες για την Ευρώπη με κρίσεις πολύ σημαντικές. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την καλή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δείξουμε ότι παρά όλες τις δυσκολίες ε, τις οποίες αντιμετωπίζει παραμένει σημαντικός παράγων για την ανάπτυξη των περιφερειών και των χωρών μας. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Όχι. Ευχαριστούμε. Αυτέ ήταν οι ερωτήσει λοιπόν και τα σχόλια από τα μέλη τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη και των Πολιτικών Ομάδων. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Προσπαθήστε να απαντήσετε αν μπορείτε. Okay, Ε, αφού έχω την ευκαιρία θα ξαναμιλήσω στα ελληνικά. Ε, θα ε, προσπαθήσω. Τέθηκαν πολλά ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για τα ερωτήματα. Δείχνω ότι και το ενδιαφέρον του Ευρωκοινοβουλίου και ειδικά της Επιτροπής Ρέτζη για την ε, Ελλάδα παραμένει πάρα πολύ ζωντανό. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο περισσότερα μπορώ από αυτά τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν. Καταρχάς, πράγματι, η συνεργασία μεταξύ των, ε, της Επιτροπής και του κράτους μέλους της Ελλάδας ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση τουλάχιστον, αλλά νομίζω αυτό ισχύει και για το σύνολο της, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι καθοριστική. Χωρίς αυτή τη συνεργασία και σε υπηρεσιακό και σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορεί να υπάρξει ε, επιτυχής υλοποίηση των προγραμμάτων και εδώ ε, θέλω να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία να εξάρω και να ευχαριστήσω και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την συνδρομή και την αποφασιστική βοήθεια που είχαμε και από την DG Regio και την Επίτροπο, την κυρία Κρέτσου, η οποία αποδείχθηκε ε, μια πολύτιμη ε, φίλη της Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θέσατε, δηλαδή ποια είναι τα μετρήσιμα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς, αυτής της προσπάθειας. Εμείς έχουμε ε, παραγγείλει αυτούς τους μήνες μια εμπειρογνωμοσύνη η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε το Σεπτέμβρη ε, μια πιο ε, μετρήσιμη ποσοτικά και ποιοτικά εικόνα για το ποια ήταν τα πραγματικά αποτελέσματα και βεβαίως αυτή θα είναι μια δουλειά την οποία θα την μοιραστούμε και με την, και με την Επιτροπή σας. Τώρα, σε σχέση με την επόμενη προγραμματική περίοδο. Και πράγματι αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα, θα πρέπει να μας απασχολεί όλους, όχι μόνο την Ελλάδα. Τι κάνουμε για το post-2020, έτσι, και επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η συζήτηση και εδώ στις Βρυξέλλες σε σχέση με την πολιτική συνοχή αλλά και το MFF, το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 είναι πάρα πολύ ζωντανή και οξία πολλές φορές νομίζω ακριβώς αυτό το οποίο είπαμε και στο, είπα και στο τέλος ομιλίας μου, ότι οι επιτυχίες της πολιτικής συνοχής είναι το καλύτερη, καλύτερη απόδειξη στην Ελλάδα, είναι η καλύτερη απόδειξη για, το, για την ανάγκη ενίσχυσης αυτής της πολιτικής και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Επειδή αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο και επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές αντίρροπες ε, δυνάμεις και εδώ στις Βρυξέλλες νομίζουμε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί αυτό το παράδειγμα για να ενισχυθούν τα επιχειρήματα υπέρ της πολιτικής συνοχή. Για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πράγματι εμείς κάναμε και μία πολιτική αν θέλετε ε, επιλογή το 2015 να ανακατευθύνουμε πόρους στο βαθμό του εφικτού και βάσει των περιορισμών του κανονισμού βεβαίω ε, σε δράσει που σχετίζονται με το κοινωνικό κράτο και δεχτήκαμε μάλιστα και κριτική γι' αυτό. Θεωρήσαμε και θεωρούμε ακόμα ότι μια από τι βασικέ συνέπειε τη κρίση ήταν η ε, η καταστροφή, αν θέλετε, πολύ σημαντικών βασικών κοινωνικών δομών και άρα η ενίσχυση προγραμμάτων που είχαν να κάνουν με την παιδεία, με την υγεία, με τι υπηρεσίε πρόνοια αποτέλεσε για εμά κεντρική προτεραιότητα και η αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ήταν καθοριστική σε αυτή την, ε, σε αυτή την ε, προσπάθεια. Και βεβαίως ε, αυτό το οποίο είπατε και το οποίο ήδη έχουμε συζητήσει με, την, με τις υπηρεσίες επιτροπής, δηλαδή πολλές φορές το overlap το οποίο υπάρχει μεταξύ προγραμμάτων ή η καλύτερη συνεργασία με μεταξύ των προγραμμάτων, εμένα θα μου επιτρέψετε όλο αυτό να το κωδικοποιήσω σε μία και μόνο λέξη. Ε, απλοποίηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί όχι εμά, απασχολεί το σύνολο των κρατών μελών. Έχει συζητηθεί πάρα πολλέ φορέ στι αντίστοιχε ε, υπουργικέ ε, συνόδου και χαίρομαι γιατί βλέπω ότι στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 υπάρχουν πολύ σημαντικέ ρυθμίσει απλοποίηση του κανονισμού που νομίζω ότι θα δώσει τη δυνατότητα για ακόμα καλύτερη αξιοποίηση όλων των προγραμμάτων. Τώρα, ε, να έρθω στα ζητήματα των μεταρρυθμίσεων, τα οποία τέθηκαν μάλιστα ε, από περισσότερους από έναν ε, ομιλητές. Πρώτα απ' όλα ε, πρέπει να πω ότι δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο παρά με τη, από, τη, με τη, διαπίστωση ότι δεν κάνουμε μεταρρυθμίσεις για τις μεταρρυθμίσεις. Κάνουμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες παράγουν πραγματικά ε, οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα για τη χώρα. Και με αυτήν την έννοια, ε, αν θέλετε και την ε, γνώμη μου, ε, ένα από τα λάθη τα οποία, πολύ βασικά δομικά λάθη τα οποία έγιναν στα ε, δύο πρώτα προγράμματα ε, προσαρμογής ήταν ακριβώς το γεγονός ότι υποτιμήθηκε η ανάγκη υλοποίησης ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων και αυτό το οποίο προκρίθηκε ήταν ακριβώς η λογική τους, της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής η οποία τελικά όπως είδαμε είχε ε, αποτελέσματα πολύ αρνητικά ε, ενίσχυση δηλαδή τα υφεσιακά φαινόμενα στην, στην ελληνική οικονομία. Με αυτή την έννοια, ε, τα τελευταία χρόνια έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες πραγματικά βοηθούν την οικονομία. Στο τρίτο πρόγραμμα έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 450 μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, έχουν να κάνουν με την υλοποίηση πολύ σημαντικών ε, προγραμμάτων τα οποία εξέλιπαν από τη χώρα για δεκαετίες. Αναφέρθηκαν ήδη κάποια από αυτά, τα ζητήματα της χωροταξίας, τα ζητήματα της απονομής δικαιοσύνης, της ηλεκτρονικοποίησης και της ψηφιοποίησης ε, υπηρεσιών ε, της δημόσιας διοίκησης. Είναι πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιήθηκαν τώρα. Επίση, να πω για μα είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο τη συνέχεια, του continuity αυτών των μεταρρυθμίσεων. Δεν, ε, η ολοκλήρωση του προγράμματο στι 20 Αυγούστου δεν σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσει οι οποίε βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίε υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με μια λογική ε, νόμων πλαισίου, framework ε, legislation δεν θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Αντιθέτω, και αυτό είναι και το νόημα και τη αναπτυξιακή στρατηγική την οποία εκπονήσαμε και καταθέσαμε και στο Eurogroup. Και επιτρέψτε μου εδώ να διαφωνήσω. Η δικιά μου πληροφόρηση είναι ότι η ανταπόκριση του Eurogroup ήταν πολύ θετική σε αυτή την πρωτοβουλία. Ε, ήταν ακριβώ αυτή. Ότι δηλαδή θα υπάρχει μια συνέχεια στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Συνέχεια όμω στην κατεύθυνση υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, οι οποίε πραγματικά ε, βοηθούν την οικονομία. Για να σα δώσω ένα, ένα παράδειγμα, ε, για να μην επεκταθώ σε, σε άλλα χωράφια, αν θέλετε, από το δικό μου χαρτοφυλάκιο. Ε, η προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει το τελευταίο 1,5 χρόνο για την απλοποίηση των διαδικασιών σύσταση και αδειοδότηση μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων, που είναι ένας νόμος πλαίσιο που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ήδη ωφελήσει περισσότερες από 32.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί με το νέο απλοποιημένο σύστημα της γνωστοποίησης μέσα σε μία μόνο μέρα, με ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή, η οποία υλοποιείται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και η οποία θα συνεχιστεί βεβαίως και το επόμενο διάστημα. Σε αυτή την προσπάθεια να πω και έχετε ε, δίκιο που το θέσατε, ότι βεβαίως αξιοποιούμε και την συνεργασία αλλά και την τεχνική υποστήριξη και βοήθεια που μπορεί να υπάρχει από, και από υπηρεσίες της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για παράδειγμα, με την SRSS έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία σε τέτοιου τύπου μεταρρυθμίσεις, όπως βεβαίως και με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΩΣΑ, ο οποίος είναι και ο τεχνικός μας σύμβουλος, ειδικά σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος. Επίσης, να πω, μιας και αναφερθήκατε στην αναπτυξιακή στρατηγική, για πρώτη φορά έχουμε μια αναπτυξιακή στρατηγική η οποία όχι απλώς περιγράφει και εδώ επίσης ε, θέλω να συμφωνήσω προτεραιότητε. Είναι πολύ σημαντικό να ιεραρχήσουμε προτεραιότητε για το ποιε μεταρρυθμίσει θέλουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Αλλά έχει και δεσμευτικό χαρακτήρα απέναντι και στου ευρωπαϊκού θεσμού, αλλά κυρίω και βεβαίω και προ την ελληνική κοινωνία. Με την έννοια ότι περιλαμβάνει ένα action plan, μια ολόκληρη λίστα δράσεων, προγραμμάτων, μεταρρυθμίσεων, ανά Υπουργείο, δεσμευτικών για αυτά τα Υπουργεία και με σαφή χρονοδιαγράμματα υλοποίησή του. Αυτό θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική ποιοτική εξέλιξη σε σχέση με το τι συνέβαινε στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Ε, έγινε μια αναφορά, και εδώ θέλω να δώσω μια διευκρίνηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου πολιτικά να είμαστε ε, σαφείς απέναντι σε αυτό. Έγινε μια αναφορά στη, στα ποσοστά ανεργία και ειδικά στην ανεργία των νέων. Πράγματι, τα ποσοστά αυτά, παρόλη τη βελτίωση των τελευταίων χρόνων, παραμένουν πάρα πολύ ψηλά. Γι' αυτό και εδώ θέλω να είμαι απολύτω σαφή. Από την δικιά μα πλευρά δεν υπάρχει καμία διάθεση και καμία λογική πανηγυρισμού για τι ε, πρόσφατε επιτυχίε για τη βελτίωση του οικονομικού κλίματο στη χώρα. Ξέρουμε ότι τα πράγματα παραμένουν πάρα πολύ δύσκολα. Θεωρούμε όμω ότι ε, οι μεγάλε δυσκολίε είναι πλέον πίσω μας ε, και αυτό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα μπροστά μας είναι σημαντικές προκλήσεις. Γι' αυτό και δεν ε, υποτιμούμε καθόλου την ανάγκη συνέχισης αυτής της ε, προσπάθειας και το επόμενο ε, διάστημα. Σε σχέση με τις ερωτήσεις που έθεσε η κυρία Σπυράκη, καλοπροαίρετα και θα απαντήσω κι εγώ καλοπροαίρετα σε αυτές τις ερωτήσεις. Καταρχάς, σε σχέση με τις δαπάνες τα νούμερα συνολικά για τις δαπάνες δείχνουν, συνολικά ενώ για την πλήρη εκτέλεση των προγραμμάτων, δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή της Ευρώπης ως προς την αξιοποίηση των πόρων του, του ΕΣΠΑ και της νέας προγραμματικής περίοδου 14-20, το γεγονός ότι αυτά τα νούμερα συνολικά ενδεχομένως είναι χαμηλότερα από αυτά τα οποία θα θέλαμε για όλη την Ευρώπη, αλλά συγκριτικά για την Ελλάδα σχέση με άλλε χώρε είναι υψηλά, δείχνει ακριβώ και την ανάγκη αλλαγή ε, βελτίωση κανονισμών, διαδικασιών, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερη απορρόφηση σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μα απασχολήσει συνολικά για την Ευρώπη και νομίζω ότι και η προσπάθεια η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή για την αλλαγή των κανονισμών, για την απλοποίηση των κανονισμών για τη νέα προγραμματική περίοδο κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί πράγματι εγώ θα πω ότι υπάρχει ένα ζήτημα Παναλαμβάνω, συνολικά όμω, για την Ελλάδα. Η Ελλάδα, ακόμα και σε αυτό το ασφικτικό περιβάλλον, αποδίδει εξαιρετικά. Ε, υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με το κατά πόσο μπορούμε να αξιοποιήσουμε του διαθέσιμου πόρου. Τώρα, σε σχέση με την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που εκεί, επιτρέψτε μου να πω, γίνεται μια, κατά τη γνώμη μα, ε, πολύ σοβαρή συστηματική προσπάθεια. Καταρχά, να πω για τι προσπάθειε τι οποίε κάνουμε εκτό ΕΣΠΑ, εκτό ε, ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με την EBRD, συμφωνίες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αποδώσει πολύ σημαντικούς πρόσθετους πόρους προς την ελληνική οικονομία, οι οποίοι δεν υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Σας υπενθυμίζω ότι μόνο για το 2017 ε, οι εκταμιεύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς την ελληνική οικονομία ανήλθαν σε ύψος ρεκόρ που ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ρεκόρ για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ακόμα για όλη την περίοδο της κρίσης και είναι πολύ σημαντική ένεση ρευστότητα στην ελληνική οικονομία. Όμως για τα ευρωπαϊκά τα προγράμματα, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά νομίζω, μια και ασχολείστε με αυτά τα θέματα, ότι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, συνιστά κρατική ενίσχυση. Ε, ε, ε υπόκειται στο καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων. Έτσι. Εκεί λοιπόν γνωρίζετε πολύ καλά ότι η χώρα μας και μόνη χώρα από τις 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλήθηκε να υλοποιήσει ένα σύστημα, πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ γραφειοκρατικό και γιατί όλο αυτό γιατί στο παρελθόν, σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρουσιάστηκαν φαινόμενα διασπάθησης πόρων τα οποία βεβαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούσε να αφήσει να συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι η προσπάθεια την οποία κάναμε για την υλοποίηση αυτού του συστήματο, για την ε, εκταμείευση αυτών των πόρων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο βάσει των περιορισμών που μα έθετε ο κανονισμό, ε, νομίζω ήταν η καλύτερη δυνατή δεδομένων ε, αυτών των συνθήκων. Και βεβαίω, μια και το ζητήσατε, θα στείλουμε και τα στοιχεία για τις εκταμιεύσεις οι οποίες έχουν γίνει αυτά τα, τα χρόνια για τη νέα προγραμματική περίοδο και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για τα νέα έργα τα οποία υλοποιούμε αυτό το διάστημα. Τέθηκε στο τέλος τέθηκαν ε, δύο πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα ε, σε σχέση με την ε, συνείδηση της βοήθειας της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης προς την Ελλάδα των πολιτών και των πολιτικών της χώρας. Έτσι. Ε, καταρχάς, εμείς συμμετέχουμε πολύ ενεργά και στην προσπάθεια η οποία γίνεται και από την DigiRigio για τα, με τα προγράμματα δημοσιότητας, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε και προς τον κόσμο, προς, την, προς τον ελληνικό λαό τις επιτυχίες αυτών των προγραμμάτων και το πόσο έχουν συμβάλει αυτά τα προγράμματα στην υλοποίηση πολύ σημαντικών έργων και δράσεων για την ελληνική οικονομία. Και υπάρχουν συγκεκριμένα κονδύλια τα οποία δαπανώνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ θα έλεγα όμω ότι πέρα από αυτό, πέρα από τα προγράμματα τη ελληνική βοήθεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ επίση η συνεργασία μα με τις αρμόδιες υπηρεσίε της Επιτροπής ε, νομίζω ότι είναι εξαιρετική. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δείξουμε ότι ακριβώς αυτή είναι η πολιτική η οποία και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη φέρνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους, ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων τα οποία πιάνουν τόπο, είναι χρήματα τα οποία βοηθούν χώρες σε κρίση όπως η Ελλάδα να εξέλθουν αυτή τη κρίση, αλλά βοηθούν και όλα τα κράτη-μέλη να καταπολεμήσουν κοινωνικές ανισότητες, περιφερειακές ανισότητες, ενδοπεριφερειακές ανισότητες και νομίζω ότι η δουλειά την οποία όλοι μας, ο καθένας από την πλευρά του και εσεί. Ε, ως ε, ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής Ρέτζη αλλά και εμείς ως μια κυβέρνηση η οποία στηρίζει ενεργά και όχι μόνο στα λόγια αλλά νομίζουμε με τις πράξεις μας την πολιτική συνοχή. Η δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να πείσουμε τους πάντε και στην Ευρώπη ότι αυτή είναι μια πολιτική η οποία πρέπει και τα επόμενα χρόνια όχι απλώς να συνεχίσει να υπάρχει, γιατί ακούσαμε διάφορα το τελευταίο διάστημα, αλλά να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, γιατί είναι μια πολιτική η οποία πατάει ακριβώς πάνω στις ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Όπως καταλάβατε, παρακολουθούμε τα έκτακτα μέτρα, τα υιοθετήσαμε για την Ελλάδα, παρακολουθούμε τα αποτελέσματα αυτών των έκτακτων μέτρων και Τώρα είχαμε αυτή την συνάντηση με ανταλλαγή απόψεων μαζί σας, που επίση είναι κάτι έκτακτο στην παράδοση των συνεδριασιών μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ήταν πολύ χρήσιμη η συνάντηση αυτή. Το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια θα συζητηθεί πάλι το θέμα. Ευχαριστούμε λοιπόν και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε, θα είμαστε σε επαφή και θα ακούμε καλά νέα από σας. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα συνεχίζουμε. Okay, we continue. Καλώς, λοιπόν, Τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θα εξετάσουμε την πρόταση κανονισμού που έχει ένα πολύ μεγάλο τίτλο. Πρόκειται για τροποποίηση λοιπόν του κανονισμού ε, περί κοινών διατάξεων όσον αφορά τις επιδόσεις ε, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κοινωνικό Ταμείο, τα διάφορα ταμεία δηλαδή κλπ. Έχουμε εδώ την κυρία Κρέλ και τον κύριο Φανίστερόι που είναι οι συγητές. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Είχαμε ήδη παλιότερα, κάναμε και ακρόαση μάλιστα για αυτό το θέμα. Και σήμερα εξετάζουμε το σχέδιο έκθεσης. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στους δύο συνεισηγητές. Ποιος από τους δύο θα αρχίσει. Παρακαλώ κύριε Φανίστεροι. Ευχαριστώ. Πράγματι είπατε κι εσείς ότι ο τίτλος είναι μεγάλος, αλλά η δουλειά γίνεται συμπυκνωμένη, έτσι. Η έκθεση είναι πολύ σύντομη, μάλιστα. Και δεν έχει εκπλήξεις, πρέπει να σας πω. Τρεις φορές έχουμε μιλήσει για την έκθεση αυτή ήδη και με τον Επίτροπο. Την τελευταία φορά συζητήσαμε πώς θα επεξεργαστούμε το θέμα εφόσον η Επιτροπή δεν μετακινείται, δεν προχωράει. Όπως είπε και η συνεισηγήτρια κυρία Κρέλ, ε, αν ε, δεν κάνει τίποτα Επιτροπή, εμεί πρέπει να κάνουμε. Ε, μιλήσαμε και με τους συντονιστές και είπαμε «Ε, ας έρθει η έκθεση, ας προχωρήσουμε γρήγορα για να είναι όλα σαφή. Αυτή είναι η πρόταση. Τώρα δεν θέλω να επαναλάβω αυτό που έχουμε πει και ξαναπεί. Η πρόταση αυτή για τις επιδόσεις δεν έχει πρόβλημα ούτε με το νομικό κείμενο, ούτε με τα ζητήματα που θέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περισσότερη ευελιξία του αποθεματικού επίδοσης να τιμήσουν τα διάφορα προγράμματα για το 2019 και μετά τα οποία έχουν καλές ε, επιδόσεις. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία κίνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περισσότερη ευελιξία, επιτάχυνση, οτιδήποτε. Ένα στόχο θέλανε και τίποτα άλλο. Και φάνηκε αυτό και στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πρώτο βήμα είναι να συμφωνήσουμε με το Ταμείο. Μετά είναι να το διευρύνουμε, να του δώσουμε νέα πνοή. Και το τρίτο βήμα πάει πιο μακριά σε αυτά τα πλαίσια. Υπάρχει πρόταση λοιπόν να απορρίψουμε Αφού δεν το αποσύρανε, εμείς θα το απορρίψουμε. Η κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Παραπέμπουμε εκ νέου ή αναπέμπουμε την έκθεση ελπίζομαι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή να μας υποστηρίξει, μία παρατήρηση. Μία χώρα μέλος είχε ενδιαφέρον για κάποιο πιλωτικό πρόγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί εάν μπορεί χωρίς αλλαγή του γενικού κανονισμού και με τις δυνατότητες που διαθέτει η Κομισιόν να μπορέσει να υλοποιηθεί το pilot project. Και οι δύο εισηγητές συμφωνούμε. Δεν συμφωνώ, ωστόσο με τι τροποποιήσεις που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Γενικό Κανονισμό. Άρα, παραπομπή εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σου μπορέσει να σκεφτεί έναν ευφυή τρόπο για να στηρίξει την Πορτογαλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. τη Τόμασιτς. Η κυρία Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει κάνει διαβουλεύσεις για την πρόταση αυτή και ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης, με τις υπηρεσίες της Κομισιόν, με την Προεδρία του Συμβουλίου και με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Και υπάρχει γενική συμφωνία ότι είναι πολύ ασθενής η στήριξη για την πρόταση. Άλλωστε, πολύ λίγοι ενδιαφερόμενοι υποστηρίζουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ συμφωνώ τα κονδύλια του Performance Reserve, του αποθεματικού επίδοσης, να δαπανώνται για έργα συνοχής. Δεν είμαι ωστόσο το ίδιο επιφλακτική όπως ορισμένοι εκ των συναδέλφων μου Ευρωβουλευτών. Συμφωνώ ότι το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να δώσει περισσότερες απαντήσεις στις ερωτήσεις που τους έχουμε υποβάλει Περισσότερε από αυτέ που έδωσε στην τελευταία συνάντηση για το πρόγραμμα αυτό και να αναλυθεί η λειτουργία του προγράμματος σε περισσότερη λεπτομέρεια. Όμω, για ορισμένε χώρε μέλη το πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει για να προχωρήσουν από μακρού αναμενόμενες διαρθρωτικές τροποποιήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Βαν μετά από την ε, κάπως θετική παρέμβαση του ECR, έχω να πω και εγώ διότι ακούσαμε τους συνεισηγητέ του Λαϊκού κόμματο και των Σοσιαλιστών Δημοκρατών και κατανοούμε εν μέρη τις προτάσεις, μάλλον του λόγου που επικαλούνται για την αναπομπή στην Επιτροπή. Ίσως να μην είναι πολύ καθαρή η πρόταση Επιτροπής, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις τις οποίες έχουμε θέσει στη διάρκεια της ακροάσεως και χρειαζόμαστε πράγματι απαντήσεις και υπάρχουν βεβαίως επιτάπητος τώρα νομοθετικές προτάσεις για το Reform Support Program για παράδειγμα. Πιστεύουμε όμως ότι η απλή, απλή απόρριψη Τη ε, προτάσεως ε, δεν είναι ο σωστός τρόπος. Διότι υπάρχουν χώρες μέλη οι οποίες σε οικειοθελή βάση θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το αποθεματικό επίδοσης για να μπορέσουν να κάνουν διαρθρωτικές μετα... μεταρρυθμίσεις. Και γιατί να τι εμποδίσουμε τις χώρες αυτές τότε να το κάνουν αυτό και ιδίως ε, όταν έχουν κάνει και διαβουλεύσεις με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως με τοπικέ τοπικές αρχές και έχουν συμφωνήσει όλοι. Για μας, την ομάδα μας, είναι η δυνατότητα να μπει ένα εργαλείο στην εργαλειοθήκη, να μην περιμένουμε άλλα δύο χρόνια μέχρι ότου υπάρξει, μέχρι ότου δημιουργηθεί μέσα στο επόμενο πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο το πρόγραμμα στήριξη των μεταρρυθμίσεων. Το ίδιο, επειδή οι λόγοι υπέρ των ε, μεταρρυθμίσεων και έχει υποστηρίξει αυτές τις μεταρρυθμίσεις και την αναγκαιότητά τους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα αυτά συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα πρέπει λοιπόν νομίζουμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία και να αρχίσουμε να επιφέρουμε καινοτομία στην πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης και μέσα σε μια οπτική βελτίωσης της θέσης μας, να έχουμε και καλύτερες δηλαδή πληροφορίες όταν θα αρχίσουμε να συζητούμε το πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων. Ως ομάδα φιλελευθέρων, Άλντε, δεν θέλουμε να αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι τώρα. Θέλουμε να επιδιώξουμε την αλλαγή. Γι' αυτό και θα καταθέσουμε επικοδομητικέ τροπολογίε που ελπίζουμε να υποστηριχτούν και από άλλε πολιτικέ ομάδε, ώστε τουλάχιστον να αρχίσουμε να συζητούμε σε τριμερεί διαλόγου με το Συμβούλιο την πρόταση αυτή και θα παρακαλέσω και του δύο συνεισηγητέ να επανεξετάσουν τη θέση του, Τουλάχιστον να κάνουμε μια δοκιμή και θα δούμε στο τριμερή διάλογο πώ μπορούμε να τροποποιήσουμε και να βελτιώσουμε τα πράγματα και να λάβουμε τι απαντήσει, στις ερωτήσει, όπω σωστά είπε και η ομάδα ECR. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ομαρζή. Ευχαριστούμε. Εμείς ε, από πλευράς μας παραμένουμε στις θέσεις μας. Όταν είχε έρθει εδώ ο κύριος Ντομπρόσκη στην Επιτροπή μας, είχαμε εκφράσει αμφιβολίες ε, σε αυτό που θεωρούσαμε παρεκτροπή, τα 21 εκατομμύρια που είχαν ληφθεί από τη συνοχή, διπλή εκτροπή ουσιαστικά διότι πήγαμε και το ψάξαμε να το βρούμε στο αποθεματικό επιδόσεων. Εμείς θέλουμε και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και το αποθεματικό επιδόσεων, οπότε θέλουμε να απορρίψουμε αυτή την πρόταση. Είναι αυτονόητο. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν άλλα σχόλια. Όχι. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Γκέλνομ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα πω δύο λόγια. Όπως ε, υπόθηκε ήδη το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απογοητευμένη από το σχέδιο εκθέσης αυτό. Αναγνωρίζω πολλά από τα σχόλια του κ. Βαν Μίλτεμπεργκ στην παρέμβασή του. Όπως είπαμε επανειλημμένος ειδικότερα όσον αφορά τις προτάσεις μας για την περίοδο μετά το 2020 για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ε, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες και στις αλλαγές και αυτή την εικόνα θα πρέπει να δίνει κιόλα. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα που έχει υποβάλει μια τροπολογία η Κομισιόν ε, στον κανονισμό κοινών διατάξεων 1420 που εισάγει προαιρετική δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να, να κάνουν χρήση αυτού παραμένει προαιρετικό. Πρέπει να συμφωνηθεί με τους εταίρους του προγράμματος, διότι μόνο έτσι μπορεί να αποδεσμευτεί ε, αυτή η χρηματοδότηση μέσω τροποποίησης υπαρχών των προγραμμάτων. Δεν είναι δηλαδή μονομερείς αποφάσεις ε, των κρατών μελών. Πρέπει να λαμβάνονται από τις διαχειριστικές επιτροπές ε, των προγραμμάτων. Τέτοιε προτάσει λοιπόν δεν πρέπει να τι βλέπουμε ω παρεκτροπή ε, εκτροπή ε, κονδυλίων. Το ακούσαμε δύο-τρει φορέ. Δεν μιλάμε για εκτροπή ε, χρηματοδότηση από το ένα μέρο στο άλλο. Οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις είναι ένα απόσπαστο κομμάτι τη συνολική οικονομική διακυβέρνηση τη Ένωση και η πολιτική συνοχή είναι ένα άλλο κομμάτι αυτή τη οικονομική διακυβέρνηση. Για να φτιάξουν λοιπόν οι μεταρρυθμίσεις μα ένα ισχυρό επενδυτικό περιβάλλον ε, μόνο έτσι μπορεί να γίνουν. Ε, η Πορτοκαλία εξέφρασε σαφές ενδιαφέρον όπως αναγνωρίστηκε να αξιοποιήσει ε, αυτή τη δυνατότητα. Από πλευράς μας είναι δυστυχίες να απορρίπτεται μια τέτοια πρόταση προαιρετική να μην μπορεί ένα κράτος μέλος να την αξιοποιήσει. Για τα όσα προτείναμε μετά το 2020 και τον τρόπο ε, εφαρμογής τους υπάρχει δυνατότητα να γίνει και ένα πρώτο βήμα για να μάθουμε παραδείγματα όπως η Πορτογαλία πάνω στα οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε πιο σταθερά τα όσα έχει προβλέψει η Κομισιόν το, μετά το 2020. Οπότε κλείνω εκφράζοντας την απογοήτευσή μας από το σχέδιο εκθέσεις αυτό. Ελπίζουμε ότι τα λόγια του ε, κύριου Βαν Μίλτεμπορ κυρίως θα εισακουστούν από την Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ κλείνει η συζήτηση. Προτείνουμε προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών για αυτή την έκθεση την 13η Ιουλίου. Τέλη της εβδομάδας, 12 ε, το μεσημέρι. εφόσον έρθουν οι τροπολογίε μέχρι τότε, θα προλάβουμε να ψηφίσουμε την εκθέση του Σεπτέμβριο, σωστά, τον Οκτώβριο. Κύριε Βαμίλτεμπορκ. Ναι, έχουμε και διακοπέ. Ε. Αν συμφωνούν οι συνεισηγητέ ε, και δεν έχει πρόβλημα η γραμματεία, θα ήθελα να μα δοθεί άλλη μια εβδομάδα για διαβουλεύσεις, Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τι τροπολογίε. Οπότε η ερώτησή μου είναι θα ήταν δυνατόν να παραταθεί η προθεσμία για την 20 Ιουλίου. Πρόεδρος βεβαίως, 20 Ιουλίου. Ευχαριστώ. Ωραία, η προθεσμία είναι 20 Ιουλίου. 12 το μεσημέρι. Καλώς, συνεχίζουμε τώρα. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για γνωμοδότηση. Γενικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό έτος 2019. Όλα τα τμήματα η υπεύθυνη επί της ουσίας επιτροπή είναι Επιτροπή Προπολογισμών. Σήμερα θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης που ετοίμασε ο εισηγητής μας, ο κύριος Βόν. Κύριε Βόν, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα έχετε διαβάσει τις προτάσεις μου, τις προτάσεις που έκανα στην γνωμοδότησή μου και θα αρχίσω με τα προφανή ότι δηλαδή η πολιτική συνοχής είναι μια από τις κύριες ε, πολιτικές μας και στην ε, πρώτη παράγραφο λέω ότι όταν στην πολιτική συνοχής επενδύουμε έχουμε 174% απόδοση σε σχέση δηλαδή με τα χρήματα τα οποία δαπανώνται στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Επίσης, στην παράγραφο 2 λέω ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πολλές φορές ξεχνάμε ότι πολλές από τις προτεραιότητές μας δεν θα είχαν υλοποιηθεί χωρίς την βοήθεια του Ταμείου Συνοχής. Στην παράγραφο 3 λέω ότι έχουμε καθυστερήσει την έναρξη του Προέδρου και οι λόγοι είναι η συμφωνία για το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Έτσι όμως καθυστερούν και άλλες συμφωνίες εταιρική σχέσης και προγράμματα με τις διάφορες χώρες μέλη και τις περιφέρειες. Πάντως θα ήταν σωστό να πούμε ότι όσον αφορά την υλοποίηση έτσι όπως την ξέρουμε τα τελευταία χρόνια και μήνες, τώρα υπάρχει κάποια επιτάχυνση που προχωράει η εκτέλεση των ε, πληρωμών. Στην έκθεσή μου επίσης λέω ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 προτείνει αύξηση 1,1% του επίπεδου των πιστώσεων πληρωμών με μείωση όμως 8,9% και 3,6% αντίστοιχα για το Ταμείο Συνοχής και την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Συνεπώς πιστεύω ότι πρέπει να εκφράσουμε την ανησυχία μας όσον αφορά τον επόμενο προπολογισμό, ότι η πρόταση αυτή δεν ανταποκρίνεται στο ρυθμό υλοποίησης των προγραμμάτων και κινδυνεύουμε να επαναλάβουμε την κατάσταση του παρελθόντος όπου είχαν συσσωρευτεί απλήρωτοι λογαριασμοί. Θα υπάρξει συνάντηση με τον κύριο εισηγητή για τον προπολογισμό και τους άλλους εισηγητές γνωμοδοτήσεων. Από ό,τι φαίνεται όλοι ζητούν περισσότερα χρήματα. Εγώ πάντως από αυτή την Επιτροπή διαφέρουμε. Γιατί αυτό που ζητάμε εμείς είναι ότι έχουν δεσμευτεί χρήματα για προγράμματα που πρέπει να πληρωθούν, οπότε τα χρήματα αυτά πρέπει να υπάρχουν στον προπολογισμό για να πληρωθούν οι λογαριασμοί. Δεν ζητάμε έτσι γενικώ παραπάνω χρήματα για να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα, όχι. ζητάμε για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς που θα μας έρθουν. Λέω και άλλα πράγματα εδώ στην γνωμοδότησή μου. Το τελευταίο που αναφέρω είναι η ερνευτική διαδικασία για την Βόρεια Ιρλανδία. Ε, ζητάω να εξακολουθήσουν τα κρατη και η Επιτροπή να στηρίζουν την ερνευτική διαδικασία και θα έχουμε βέβαια και έκθεση πρωτοβουλία όσον αφορά ε, τα χρηματοδοτικά προγράμματα στη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Πάντως υπάρχει χρηματοδότηση και πρέπει να συνεχιστεί και να γίνει τώρα, να μην καθυστερήσει, αλλά να συνεχιστεί βέβαια και μετά το 2020, ό,τι και να γίνει τότε. Αυτά είναι τα σχόλιά μου για την έκθεσή μου. Προσβλέπω στα σχόλια των συναδέρφων και τροπολογίε στη γνωμοδότηση αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Οι σκιώδεις εισηγητές έχουν τώρα το λόγο. Ε, εκ μέρους του κύριου Ντόιτς κάποιο. Ναι, δεν τον είδα εδώ τον κύριο Ντόιτς, λέει ο κύριος Φανίστεροι. Οπότε εγώ μπορώ να πω κάτι εκ μέρου του ΕΛΚΑ. θα σκεφτόμουν για το 2019, νέτο μεταρρυθμίσεων. Ε. Είχαμε συζήτηση και όντως το 2019 είναι που αρχίζουμε ε, αυτή την νέα περίοδο και θα έπρεπε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις διαδικασίες. Ευχαριστούμε κυρία Τόμασιτς. Σας ευχαριστώ. Στηρίζω τη γνωμοδότηση γιατί υπογραμμίζει πόσο μεγάλη σημασία έχει η πολιτική συνοχή, ότι είναι βασική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθάει να μειωθούν οι κοινωνικές, οικονομικές ε, και άλλες διαφορέ στι διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες, ε, βοηθάει και ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη, την ύπεθρο και ενθαρρύνει ώστε να προχωρήσουμε και σε νέες περιβαλλοντικές επιλογές για λιγότερο άνθρακα. Ε, πρόκειται για μία απόδοση της τάξης του 174%. Λιγότερες επενδύσεις σημαίνει λιγότερη ανάπτυξη και λιγότερη απασχόληση για τους πολίτες. Θέλουμε να συνεχίσουν τα κονδύλια συνοχής, να εξακολουθούν να παίζουν το ρόλο που έπαιζαν μέχρι σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιπλέον θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία για να πετύχουμε τι κύριε προτεραιότητε που περιλαμβάνονται και στο σχέδιο προπολογισμού για το 2019. Δηλαδή να έχουμε μια ευρωπαϊκή οικονομία με περισσότερη αντοχή, περισσότερη αλληλεγγύη και ασφάλεια όχι μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτής και έτσι μόνο θα μπορέσει να υλοποιηθεί ικανοποιητικά ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κατάνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, συναδελφό τον κύριο για τις ε, πολύ καλές προσπάθειες που έκανε για αυτή τη γνωμοδότηση. Το σχέδιο αυτό εξετάζει πολύ επιτυχημένα την πολιτική συνοχή, ίσως την πιο σημαντική και επιτυχημένη πολιτική και τα ε, θετικά της αποτελέσματα. Όπως ε, έχει το πρόγραμμα σήμερα, ε, η εκθέση περιγράφει ότι η υλοποίηση έχει μπει στη σωστή ταχύτητα, ότι εφαρμόζεται πολύ σωστά, σημαίνει ότι τα κονδύλια ε, έχουν προσαρμοστεί σε πραγματικές ανάγκες των κρατών μελών. Παρά αυτό, σε ορισμένες χώρες ε, είναι πολύ αισιόδοξε οι προβλέψεις γιατί με τις πραγματικές ανάγκες και τις εκτιμήσεις. Οπότε, εγώ δεν θα ανησυχούσα ε, τόσο πολύ για τις εκτιμήσεις της Επιτροπής. Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι παραπάνω για την προβολή του προϋπολογισμού για το πόσο ορατό είναι. Θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για τι επενδυτικέ δυνατότητε των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Να αναφέρουμε του στόχου και τα καλά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί. Συνολικά χρειαζόμαστε πιστεύω έναν προπολογισμό πιο ορατό, πιο αποτελεσματικό που να αντιμετωπίζει τι σημερινέ και ρεαλιστικές ανάγκες των πολιτών μα και των κρατών μελών μα. Αυτό πιστεύω πρέπει να υπογραμμίζεται στο κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάρζε. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω πόσο υψηλής ποιότητας είναι η έκθεση αυτή του κρυβών. Συμφωνώ με το σύνολο των θεμάτων που τέθηκαν. Ήθελα απλά να υπογραμμίσω ότι από πλευράς μας θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να αναφέρεται πιο σαφώς η δική μας θέση όσον αφορά το θέμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Και πράγματι πολύ σωστά υπενθυμίσατε ότι του χρόνου θα έχουμε το αποθεματικό επιδόσεων. Οπότε να επιμένουμε παραπάνω σε αυτό. Χαιρόμαστε για το σημείο που αφορά την Βόρεια Ιρλανδία και τη διατήρηση της ειρήνης. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό για την ομάδα μας. Τέλος, πιστεύω ότι καλό θα ήταν να υπενθυμίσουμε ε, ποιες είναι οι νέες πολιτικές που χρηματοδοτεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες θα αποδυναμώσουν την πολιτική συνοχή. Αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στην αμυντική πολιτική και εν ώψη του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Πάντα καλό είναι να υπενθυμίζουμε ότι οι νέε προτεραιότητε, ε, μεταναστευτική πολιτική, ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας άμυνας θα αποδυναμώσουν την πολιτική συνοχή. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω τους άλλους κοιόδες. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Όχι. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω την έκθεση αυτή σε αντίθεση με τα προηγούμενα μου σχόλια. Ένα-δυο σχόλια είχα. Σημειώνουμε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν ειδικότερα για το σημείο 4, αλλά από την πλευρά τη Κομισιόν θεωρούμε ότι το επίπεδο των ε, κονδυλίων είναι επαρκές ε, για να καλύψει το σημερινό ρυθμό υλοποίησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα σχόλια στο σημείο 5 όσον αφορά τον καθορισμό, το χαρακτηρισμό. Η Κομισιόν εργάζεται, συνεργάζεται στενά με τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα ε, οριστικοποιήσει την θέση ορισμού τους, οπότε η θέση του Κοινοβουλίου εκεί είναι σημαντική, διότι έχουμε συμφωνήσει ότι το να μην έχουμε ακόμα ορίσει αρχές ε, στα μέσα του 2018 είναι απαράδεκτη κατάσταση. Ε, δείχνει ε, υποαρνητική δίνει αρνητική εικόνα σε κάποιες πτυχές της πολιτικής συνοχής. Και τέλος θα ήθελα να υποστηρίξω πλήρως τα όσα λέει ο εισηγητής στο σημείο 7 όσον αφορά το πρόγραμμα της Κομισιόν η οποία θα συνεχίσει όπως έκανε στο παρελθόν να υποστηρίζει το πρόγραμμα PIS ε, ε, και τη διαδικασία, την ειρηνευτική διαδικασία, διαδικασία στην Βόρεια Ιρλανδία. Ευχαριστούμε κύριε Βόν, εκτός μικροφώνου. Εκτός μικροφώνου. Αισθάνομαι αδύναμο σήμερα το πρωί, λέει ο κύριο ομιλητής. Δεν σε το κουμπί αρκετά. Για τα όσα είπε η Κομισιόν και όσα είπαν και οι συνάδελφοι, υποστηρίζω τον κύριο Βανίστερο και τον κύριο Μαζέ που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 6 που αναφέρεται στο SRSP. Θα μπορούσαμε εκεί να αλλάξουμε λίγο τη διατύπωση με κάποια τροπολογία ενδεχομένως και με μεγάλη μου χαρά και εγώ να το δούμε αυτό το πρόγραμμα στήριξης διευθυντικών μεταρρυθμίσεων αναφέρθηκα η... το πως ε, τι, τι επιδρασία έχει η πολιτική συνοχής και τα νέα ταμεία, πώς θα, τα, πώς θα επηρεάσουν την πολιτική συνοχή. Ε, ε, θα πρέπει να κάνουμε μια τροπολογία γι' αυτό. Και το τελευταίο που θέλω να πω ήταν αυτό που είπε η κυρία Καταρίν για την προβολή των Ευρωπαϊκών Ταμείων είναι κάτι που έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην Επιτροπή μας. Και όταν πηγαίνουμε ως αντιπροσωπεία σε διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντα εκεί επισημαίνουμε ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και ότι ο κόσμος πρέπει να αντιλαμβάνεται πώς συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τόσο σημαντικά έργα. Είναι κάτι το οποίο υποστηρίζω ολόψυχα και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. προτινόμενη ημερομηνία για τις τροπολογίες 3η 17 Ιουλίου 12 το μεσημέρι. Δεν θα έχουν αντίρρηση πιστεύω οι σκιώδεις και όλοι οι υπόλοιποι. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία λοιπόν προθεσμία 3η 17 12 το μεσημέρι και έτσι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην συνεδρία του Σεπτεμβρίου. Ωραία. Τελειώσαμε με αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Και δίνουμε τώρα το λόγο στον κύριο Ομαρζέ να μας παρουσιάσει την ενημέρωση σχετικά με την ε, αποστολή μας ε, στην Βοστόνη και την Ουάσιγκτον. Έχετε το λόγο κύριο Ομαρζέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή μας Περιφερειακής Ανάπτυξης όντως ε, πήγε 7 με 11 Μαΐου στην Ουάσιγκτον και στη Βοστόνη. Πρόεδρε εγώ. Το θέμα μας ήταν η ανάπτυξη στρατηγικών εφίους ειδίκευσης, καινοτομία, έρευνα στα πλαίσια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στι ΗΠΑ. Πρέπει να σας πω ευθύ αμέσω ότι στο σύστημα οργάνωσης των ΗΠΑ δεν βρήκαμε το αντίστοιχο της πολιτικής συνοχής έτσι όπως τη γνωρίζουμε εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το λέω ευθύ εξ αρχής. Στην Ουάσιγκτον συναντηθήκαμε με μέλη από το κογκρέσο εκεί και μιλήσαμε και για φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, συναντηθήκαμε με δύο διοικητικούς οργανισμούς της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης που ασχολείται με την οικονομική οργάνωση και ένα τμήμα του εμπορικού επιμελητηρίου κατά κάποιο τρόπο, Business Administration, που είναι μια αμερικανική κυβερνητική οργάνωση με την οποία συζητήσαμε το θέμα της καινοτομίας, των περιφερειακών προγραμμάτων ε, στρατηγικής καινοτομίας ε, και για τις επιχειρήσεις. Στην ε, Βοστόνη που πήγαμε διαπιστώσαμε όντως ε, πρόκειται για πολιτεία ε, που βρίσκεται σε εχμή όσον αφορά την ε, έρευνα και την κοινοτομία. Στη Βοστόνη υπάρχουν πανεπιστήμια υψηλού επίπεδου που επισκεφθήκαμε το MIT και το Harvard που όπως το ξέρετε βρίσκονται μεταξύ των πρώτων πανεπιστημίων ανά τον κόσμο. Στο MIT ανταλλάξαμε απόψεις για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίζουν οι πόλεις στο μέλλον εξαιτίας της δημογραφικής εξέλιξης και της κλιματικής αλλαγής. Συζητήσαμε επίσης να δούμε το big data, τι απαντήσεις μπορεί να δώσει στην ανάπτυξη των πόλεων. Και αναφερθήκαμε και στις νέες θαλάσσιες οδούς. Στο ΕΜΕΤΗ συζητήσαμε και περί τεχνητής νοημοσύνης. Τι, ποιοι είναι οι προβληματισμοί. Αλλά δεν θα πω σε λεπτομέρειες στο Χάρβερτ Συζητήσαμε με το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών για τις ανταλλαγές με την Ευρώπη για το πρόγραμμα Horizon 2020 και επισκεφθήκαμε και διάφορα προγράμματα όπως είναι το zero, δηλαδή πρόκειται για μηδενική, το house zero, για μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Ήμασταν προσανατολισμένοι κυρίως στα θέματα της έρευνας και της καινοτομίας. Πάντως δεν μπορέσαμε να ασχοληθούμε με τις δαφικές διαφορές ή τις ανισότητες, τις κοινωνικές οι ερωτήσεις που θέσαμε σχετικά με αυτά τα θέματα έμειναν λίγο πολύ αναπάντητες. Από την άλλη όμως, για ό,τι έχει να κάνει με τα αποτελέσματα των ε, πολιτικών σε θελοντική βάση για την έρευνα και την καινοτομία, από εκεί είχαμε πολλά να μάθουμε. Και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν και αντίστοιχα μοντέλα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα η αποστολή αυτή. Ευχαριστώ το προσωπικό που συνεισέφερε κατά πολύ στην επιτυχία της αποστολής αυτής και θέλω και να υπογραμμίσω τη συνοχή και την ποιότητα συνοχής που διαπιστώθηκε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Το τελευταίο σχόλιο ήθελα να πω, αλλά είναι και ο κύριος Βανίστερ Ρόι. Σας ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας για την έκθεση. Πρώτα συναντηθήκαμε με τους Ευρωπαίους πρέσβεις και η πρώτη ερώτηση ήταν μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο πρέσβης μας απάντησε δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, μπορείτε να πάτε σπίτια σας. Είπε εδώ υπάρχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση κινούμεθα μέσω της φορολογίας, ζωνών ανάπτυξης δημοσιονομικών μέτρων με τα οποία λειτουργεί η οικονομία. Δεν ρίχνουμε λεφτά στις χώρες όπως γίνεται εδώ στην Ευρώπη. Επιτρέπουμε την εισρωή κονδυλίων και οι πολιτείες έχουν τη δική τους πολιτική για την ανάπτυξη. δεν πάμε σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Βοστόνη να πούμε να αυτό είναι και αυτό το, το επόμενο βήμα. Συχνά συνεργάζονται με πανεπιστήμια, αλλά δεν βάζουν λεφτά. Δημιουργούν τις συνθήκες για να αναπτυχθεί η οικονομία, αλλά είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση στη συνοχή. Όπως είπε και ο κύριος Ομαρζή. Δεν υπάρχει αντιστοιχεία, δεν υπάρχει αντίστοιχο, δεν υπάρχει ισοδύναμο με αυτό που έχουμε εδώ ως πολιτική συνοχής και στην καινοτομία ε, πράγματι έχουμε τόσα μάθημα από αυτού. τεχνητή νοημοσύνη. Είδα πράγματα που δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Βεβαίω έχω και του δικού μου περιορισμού. Αλλά εκεί ε, ε, γεννιέται η νέα γενιά τη τεχνολογία, Εκεί επινοείται, εκεί εφευρίσκεται. Ήταν πολύ καλή ιδέα που πήγαμε. Δεν βλέπω τον κύριο Μίλτενμπεργκ που σίγουρα θα ήθελα να σχολιάσει και δική του ιδέα ήταν να, πάμε. Πάντω επιτυχής αποστολή. Αυτό οφείλω να πω. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βανίστελροϊ. Άλλος κανεί. Σήμερα μιλούμε βέβαια για ε, ειδικέ αποστολέ. Ευχαριστώ τον κύριο Μαρζέ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση της αποστολής στι ΗΠΑ, στη Βοστόνη. Εδώ ολοκληρώνεται η, η ημερήσια διάταξη της ε, σημερινή μα συνεδρίαση, του πρωινού δηλαδή. Έχω τώρα ερώτηση για του συντονιστέ. Μπορούμε να συνεχίσουμε συνεδρίαση των συντονιστών τώρα αμέσω. Αυτή την ερώτηση απευθύνω και στου συμβούλου πολιτική. Μπορούμε να συνεχίσουμε με την συνάντηση των συντονιστών ή θα πρέπει να διακόψουμε και να επαναλάβουμε στις 12 όπως είχε αρχήθεν σχεδιαστεί. Πεςτε μου, πέντε λεπτά θέλετε οι ε, σύμβουλοι πολιτικής, policy advisors, μπορούμε να διακόψουμε για πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά. Ωραία λοιπόν, πέντε λεπτά και συνεχίζουμε με τους συντονιστές.